Τώρα η εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα ε, θεσμικά όργανα. Είναι το τέλος της αρχής, θα έλεγα. Ε, ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό. Θα ψηφίσουμε αύριο στις 11.30. Θα προχωρήσουμε λοιπόν με την επόμενη έκθεση, την έκθεση του κυρίου Όουσκι, ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων. Δίνω το λόγο στον εισηγητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην έκθεση αυτή ο στόχος μας είναι να προστατεύσουμε περισσότερο και καλύτερα το κοινό και την υγεία του. Λόγω του αρνητικού αντικτύπου που έχει ο θόρυβος στην υγεία κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ιατρικός. Είναι θέμα λιλικίας λοιπόν και θα πρέπει να υπάρξει προστασία. Η Επιτροπή εστιάζει την προσοχή της μόνο στα επίπεδα θορύβου των φορτηγών και των μηχανοκίνητων οχημάτων. Η βάρος του συνόλου της έκθεσης, εγώ ήθελα να είμαι πολύ πιο περιεκτικό στο κείμενό μου εξ αρχής. Είμαι πεπισμένος ότι η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να ε, περιλαμβάνει και ε, την επιφάνεια των ε, δρόμων, το δόστρωμα, την ασφαλτόστρωση, την ποιότητα των ελαστικών, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν το θόρυβο. Τρία βασικά ζητήματα έχουν αναδεθεί. Έχουμε την ετικετοθεσία, τη σήμανση, την υποχρεωτική δήλωση των ε, επιπέδων θορύβου, το σύστημα AVAS που είναι το σύστημα approach and vehicle audible systems, δηλαδή συστήματα που ε, βγάζουν ήχους για να προειδοποιήσουν για ένα όχημα που πλησιάζει. Όλα αυτά θα πρέπει να τα περιλάβουμε λοιπόν ε, στην νομοθεσία μας. Νομίζω ότι έχει βρεθεί λύση για τα πρώτα δύο σημεία. Υπάρχει συνένεση από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ε, το σημείο τριβής ήταν το παράρτημα 3 και επικράτησε η άποψη ε, των σοσιαλιστών. Οφείλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ε, γίνεται μια εκστρατεία αρνητική κατά της έκθεσης αυτή στην Επιτροπή ε, με επικεφαλή σε μια οργάνωση από τις κάτω χώρες και δυστυχώς τη στήριξαν αυτή την εκστρατεία διάφοροι συνάδελφοι. Ε, θέλησαν να με παρουσιάσουν ως εκπρόσωπο και μισθωτό της αυτοκινητοβιομηχανίας τελικά. Ε, δυσφήμισαν το όνομά μου και αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτό το εγχείρημα δημιούργησαν μια ψεύτικη ιστοσελίδα η οποία υποτίθεται αποδεικνύει τις, τους δεσμούς μου με την αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι κατάφορα ψέματα όλα αυτά. Ε, όμως ε, τα έχουν πιάσει τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τα διαδίδουν και αυτό έχει επισκιάσει τη δουλειά που έχει γίνει στην Επιτροπή μας τις τελευταίες εβδομάδες. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ματίας Κρότε, ο οποίος έκανε μια ξεκάθαρη δήλωση που απέκλεισε ε, μεροληψία σε βάρος μου και μεροληψία από πλευράς μου, σε σχέση με αυτό βέβαια. Τελικά, ως προς το παράρτημα 3, το οποίο προτείνω, θεωρώ ότι είναι μια πραγματικά καλή συμβαστική λύση που μειώνει τα επίπεδα θορύβου των μηχανοκίνητων οχημάτων και από την άλλη επιτρέπει στην αυτοκινητοβιομηχανία να διαχειριστεί αυτό το τεχνικό δύσκολο προαπαιτούμενο. Πρέπει να πούμε ότι δεν εξετάζουμε μόνο τον αντίκτυπο στην υγεία μας, αλλά εξετάζουμε και τον αντίκτυπο των αποφάσεων μας σε 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Είναι οι άμεσα και έμεσα απασχολούμενοι στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αν θέλουμε βιώσιμη λύση θα πρέπει να υποψηφίσουμε την τροπολογία υπαριθμών 61. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε τη συζήτηση να ακούσουμε τον Επίτροπο. Κύριε Ταγιάννη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κύριο Ότσχη, τους κοιόδης συζητητές και την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, για το έργο τους. Η πρόκληση, η πραγματική πρόκληση αυτής της πρότασης είναι πώς θα βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ τριών αξώνων τα περιβαλλοντικά στοιχεία, το κόστος ε, και το χρόνο για την βιομηχανία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι οι διάφορες αυτές ανησυχίες ε, αποτέλεσαν ε, αντικείμενο δύσκολων συζητήσεων εντός του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του κειμένου, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Η πρόταση θέλει καταρχάς να διασφαλίσει ότι θα έχουμε μία πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά, να προστατεύσουμε το περιβάλλον ε, για τους πολίτες μας και να προάγουμε την ανταγωνιστικότητα των οικονομικών φορέων. Δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε κανέναν από αυτούς τους στόχους, οι οποίοι είναι αλληλένδετοι μάλιστα, ιδίως εν καιρό οικονομικών δυσκολιών για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει παρόλα αυτά να θυμηθούμε ποιο είναι το πλαίσιο της πρότασης. Πάνω από το 50% του πληθυσμού της Ένωσης εκτίθεται σε θορύβους οι οποίοι θεωρούνται απαράδεκτοι από τους επιστήμονες και τους ε, ειδικού στον τομέα της υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανέλαβε ότι η υπερβολική έκθεση στο θόρυβο αποτελεί παράγοντα άγχος, καρδιακών παθήσεων και αϊπνίας. Και για να καταπολεμήσουμε του θορύβου στου δρόμου, θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, θα πρέπει να παρέμβουμε στις οδικέ υποδομές, στους κανόνες κυκλοφορίες, στου ελέγχου τη αστυνομία, στην ενημέρωση των οδηγών και τέλο στα χαρακτηριστικά των οχημάτων. Και θα πρέπει να εκπονήσουμε τεχνικού κανόνε για τα οχήματα που σημαίνει ότι θα πάμε στη ρίζα του προβλήματο. Γι' αυτό ακριβώ έχουμε και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το θόρυβο των οχημάτων από το 1970. Σχεδόν 45 χρόνια δηλαδή και τα όρια ε, το, συγχωρήπανσης τροποποιήθηκε, το, τροποποιήθηκαν το 1995. Κατόπιν όμως διαπιστώθηκε ότι παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν τα ανώτατα όρια, δεν ε, μειώθηκε η χορύπανση όσο περιμέναμε ως ένα έθιο ήταν το γεγονός ότι δεν είναι ανταπροσωπευτικό των εκπομπών ε, των ε, οχημάτων. Γι' αυτό ακριβώς προτάθηκε να έχουμε ένα νέο στοιχείο το οποίο είναι πιο αντιπροσωπευτικό. Πρόκειται για ένα επίπεδο το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς, το ετοίμασε η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για το θόρυβο των οχημάτων και εκεί συμμετέχουν και οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών ε, επιβεβαιώθηκε, επαληθεύθηκε για τρία χρόνια με ε, βάση δοκιμές σε αυτοκίνητα οχήματο και προβλέπεται να μειωθούν τα ανώτατα όρια θορύβου σε δύο στάδια σε πρώτο στάδιο δύο χρόνια μετά την έγκριση της πρότασης για να προσαρμοστούν τα παρόντα όρια στη νέα μέθοδο υπολογισμού. Και το δεύτερο στάδιο είναι πιο σημαντικό και θα πρέπει να γίνουν και αλλαγέ στα οχήματα. Θα εφαρμοστεί 5 με 7 χρόνια ε, μετά την έγκριση της νομοθετικής πράξης. Προτείνεται να μειωθεί ε, το επίπεδο θορύβου κατά 4 δεσιμπέλ για τα ε, ελαφρά οχήματα και κατά 3 δεσιμπέλ για τα βαρέα οχήματα. Μειώνεται έτσι πολύ, κατά πολύ ο αριθμός των ατόμων που πλήττονται από την ηχορύπανση, ε, αν εγκριθεί η πρόταση, και σύμφωνα με την αξιολόγηση επιπτώσεων είναι πολύ σημαντικά τα ωφέλη, 20 πλάσια μάλιστα για την κοινωνία, σε σχέση με το τι θα επιβάλλουμε στον ε, κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ευχαριστώ την Επιτροπή Περιβάλλοντος και ελπίζω ε, να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα μιλώ σε αυτή την προκεχωρημένη ώρα εξ ονόματος της συναδέλφου Άνια Βάισμπεργκερ που είναι ε, αρμόδια για την γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και Προστασίας των Καταναλωτών. Είναι σημαντική αυτή η πρόταση για τη μείωση της ε, η χορύπαση, ε, αλλά έχει να κάνει και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την επιλογή ε, του οχήματος όταν αγοράζει κανείς αυτοκίνητο. Η τυφλή. Ε, ε, τα παιδιά, οι ποδηλάτες και οι πεζοί έχουν πρόβλημα ε, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτροκίνητα τα οποία είναι αθόρυβα. Γι' αυτό και το σύστημα AVAS προτείνεται ένα προειδοποιητικό με ήχους, με ψιθύρους και θα πρέπει οι εταιρείε να προσαρμόζονται για να είναι ακριβώς εύκολο να καταλάβει κανείς τι είναι αυτό το όχημα που έρχεται και να κάνει ε, αντίστοιχο θόρυβο με ένα συμβατικό. Να είναι προειδοποιητικό αυτό ο ήχος. Ε, η προστασία των καταναλωτών είναι σημαντική και η Επιτροπή μας ε, προτείνει να υπάρχει ένα σήμα που να ενημερώνει του πολίτε όταν θέλουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο οι καταναλωτές για τι εκπομπέ θορύβου και τα επίπεδά Του Ευχαριστώ για τρία λεπτά ο κύριο Παρνιό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Όσο εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής ε, Μεταφορών και Τουρισμού, καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των επίπεδων θορύβου των μηχανοκίνητων οχημάτων. Τα στοιχεία είναι από την ΠΟΑΗ. Το 2% των καρδιακών κρίσεων στην Ευρώπη οφείλεται ε, σε ε, θορύβους άνω των 60 δεσιμπέλ. Ο θόρυβος από τους σιδηροδρόμους αλλά και από τους δρόμους ε, είναι και η πηγή, αν θέλετε, η αιτία 50.000 ε, καρδιακών προσβολών και 200.000 ε, καρδιακιακών παθήσεων. Αυτά είναι τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και τα, τους κανόνες τους έχουμε από το 96 πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθούν και να μεταρρυθμιστούν. Εμείς θελήσαμε να συμπληρώσουμε την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής να έχουμε μια ενιαία προσέγγιση υποχρέωση ε, ύπαρξης ενός ελάχιστου θορύβου για τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα και την προώθηση αυτού του συστήματος ε, ηχητικής προειδοποίησης. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ρεαλιστικούς αλλά και εφικτούς στόχους και γι' αυτό η γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών προτείνει την υιοθέτηση νέων ανώτατων ορίων και μάλιστα σε βάθος χρόνου θέλουμε να μειώσουμε ε, κατά 4 δεσιμπέλ σε 8 χρόνια 2 δεσιμπέλ μετά από, 20, μετά από 6 χρόνια και τελικά όλα αυτά να αφορούν το σύνολο των οχημάτων που θα διατίθενται στην αγορά. Αυτή είναι μια συμβιβαστική λύση που έχει επιτευχθεί με το ΕΛΚ, σε συνεργασία με το ΕΛΚ, έτυχε μεγάλη στήριξη στην Επιτροπή και ελπίζω και πιστεύω ότι την τροπολογία αυτή τη συμβαστική την συμπεριέλαβε συνάδελφος Ζούντιτ Περκές ε, εξ ονόματος της ΓΚΟΕ, των Πρασίνων και του Άλντε. Στην κρίση λοιπόν αυτή τη στιγμή ε, που βιώνει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είναι σημαντικό οι κατασκευαστές να έχουν επαρκή προθεσμία για να, αρκετή προθεσμία για να ε, τηρήσουν τις νέες ευρωπαϊκές δεσμεύσεις. Σίγουρα οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές είναι θετικός διακείμενοι προκειμένου να μειωθεί ο θόρυβος των μηχανοκίνητων οχημάτων. Αυτή η μείωση λοιπόν του θορύβου θα πρέπει να γίνει αλλά να γίνει ρεαλιστικά, με εφικτό τρόπο, χωρίς να διατηρηθούν οι οικονομικές ισορροπίες στη σημερινή περίοδο κρίσης στην Ευρώπη. Και η τροπολογία της κυρίας Μαρκές είναι μια πολύ καλή συμβαστική τροπολογία. Είναι πολύ ε, πιο ε, ευέλικτη σε σχέση με τα προτινόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κλάδος θα μπορέσει να αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία για να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους σε λογικές προθεσμίες. Μιλούμε για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή στρατηγική η οποία ε, θα πρέπει να ε, κάνει όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους ως προς την έρευνα ε, για τα οχήματα ε, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτά ήθελα να σας μεταφέρω εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστώ κύριε ο κύριο Σταταρέλα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αντιαμφισβήτητο ότι πρέπει να εγκρίνουμε αυτή τη δέσμη νομοθετικών μέτρων. Συμφωνούμε όλοι ως προς το στόχο. Η διαφορά είναι ο τρόπος, ο χρόνος και η τεχνολογία. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναφέρθηκε και από κάποιον άλλον σήμερα. Εδώ και αρκετό καιρό μας λέει ότι πρέπει να παρέμβουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα, διότι ο θόρυβος, ιδίως στις μεγάλες πόλεις, επί δρά ε, στην ε, υγεία των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε την υγεία των πολιτών μας, να βελτιώσουμε το βιωτικό τους επίπεδο και να μειώσουμε τα ντεσιμπέλ τα οποία οδηγούν, οδηγούν σε άγχος και ασθένειες. Αλλά δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να δολοφονήσουμε τον, ε, την αυτοκινητοβιομηχανία. Ιδίω αυτή τη στιγμή που η αυτοκινητοβιομηχανία βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Ο θόρυβος είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων. Δεν προκύπτει μόνο από τα αυτοκίνητα, αλλά και από το θόρυβο των υποδομών στις πόλεις. Ε, στις πόλεις δε συνεισφέρει ακόμα περισσότερο. Δεν θα πρέπει να τα ρίχνουμε όλα στα αυτοκίνητα. Και το λέω αυτό κυρίως στους συναδέλφους της αριστεράς και τους σοσιαλιστές, ε, οι οποίοι δικαίως ε, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα θέματα της αποσχόλησης η πτώση του ε, αυτοκινητοβιομηχανίας δεν έχει συνέπειες μόνο για την τιμή των αυτοκινήτων, μειώνει και την, το επίπεδο απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και την πτυχή αυτή. Η ουσία όλης αυτής της νομοθεσίας η οποία είναι πολύ τεχνικής φύσεως και μάλλον δεν ενδιαφέρει και ιδιαίτερα τους συναδέλφους. Το συζητήσαμε ελάχιστα στην ε, ε, Επιτροπή ε, περιορίζεται στις τροπολογίες 51 και 61. Να υπενθυμίσω ότι 51 πέρασε με διαφορά μία ψήφου και μόνον και είναι ε, ουτοπικό να οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να απορρίψουμε την 51 και να την καταστήσουμε με την 61. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά η κυρία Μερκής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε. Κάθε ψήφος μετράει από ό,τι ξέρω και αυτό αύριο θα ισχύσει. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς ο θόρυβος είναι από ό,τι φαίνεται τα μεγαλύτερα προβλήματα στην υγεία. 50.000 περίπου καρδιακές προσβολές ε, συνδέονται άμεσα ε, από ενοχλήσεις ε, λόγω θορύβου. Και αυτό είναι κυρίως άνθρωποι με χαμηλών εισοδημάτων που ζουν κοντά σε αυτοκινητοδρόμους, σε κέντρα πόλεων με κακή χωρί, μόνωση και εκτεθειμένοι στο θόρυβο. Και τώρα πώς το σταθμίζουμε αυτό απέναντι στις θέσεις απασχόληση. Θα επανέλθω στη συνέχεια. Πώς λύνουμε σήμερα ε, το πρόβλημα του θορύβου. Αντιμετωπίζουμε στα συμπτώματα. Σε όλη την Ευρώπη ε, ε, φτιάχνουμε υποδομές, μεγάλους τείχους, προστατευτικά για το θόρυβο πολλές φορές από τα διαρθρωτικά ταμεία. Και ποιος θέει το αυτοκίνητο. 60 ε, ε, ευρώ αναγιώταχή και 750 ευρώ ε, αναφορτηγό κοστίζει η μετατροπή. Και συζητούμε για την καινοτομία, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι τα εννοούμε όλα αυτά. Κύριε Επίτροπε, δεν ισχύει αυτό και μπορείτε να το πείτε και στους ομολόγους σας. Ε, υπάρχουν ε, ε, μελέτες σκοπιμότητας που δείχνουν ότι θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, δεν θα χαθούν με αυτό τον κανόνα εάν ε, εφαρμοστεί σωστά. Θα μειωθεί και το κόστος των συστημάτων υγείας και κυρίως θα αυξηθεί η υγεία για όλους τους Ευρωπαίους. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά τώρα ο κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Εδώ και ένα χρόνο τώρα συζητάμε αυτή την νομοθεσία. Γιατί διαρκεί τόσο καιρό. Και εγώ εκπλήσωμαι που δεν το είπε κανένας προαλλαλής σας. Είναι κακή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκανε πρόταση νομοθετικού κειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν ανταποκρίνεται στις ίδιες τις απαιτήσει τους για την νομοθεσία. Ε, η καρδιά της ε, νομοθεσίας είναι το παράρτημα 3 με παλιά στοιχεία για τα οχήματα της δεκαετίας του 80 και εμείς καλούμεθα να το διορθώσουμε. Πώς ορίζονται ε, οι κατηγορίες αυτοκινήτων με, με μα εδώ χρειάζονται φυσική και μάλιστα με ειδικότητα της φυσικής, ακουστική για να δώσουν αποτέλεσμα. Η συζήτηση που έγινε στο Κοινοβούλιο δεν ήταν κάτι που πριτάνευε πάντα η λογική. Δεν μπορούμε να ζητάμε για γιοταχή ε, επίπεδα θορύβου από τη μια ε, που ανταποκρίνονται σε ηλεκτροκίνητα οχήματα και από την άλλη να ζητάμε και ελάχιστο θόρυβο για τα ηλεκτροκίνητα γιατί ε, το αθόρυβο μπορεί να είναι και μουγκό τελικά. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνουμε με τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Η ιδεολογία ε, έχει παρισφρήσει τόσο πολύ που είναι παράλογα αυτά. Ε, θα πρέπει να συζητήσουμε, ε, λέτε, για τα αθλητικά τα αγωνιστικά μάλλον ε, αυτοκίνητα. Μα τι ανοησίες είναι αυτές οι ιδεολογικές. Είναι κάτω από 1% των οχημάτων αυτών ε, τα μηχανοκίνητα, του, του μηχανοκίνητου ε, αθλητισμού. δεν είναι καλή η πρόταση για τον κανονισμό. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να πάρει απόφαση με υπευθυνότητα και μιλώ για το σχέδιο τροπολογίας 62 που είναι συμβιβαστική. Θα πρέπει να ε, πάμε σε αξιόπιστες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία. Για δύο μισή λεπτά η κυρία Χάση. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα σε μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες στη Φιλανδία ένα άρθρο έγραφε ότι μισό εκατομμύριο Φιλανδοί υποφέρουν από τον ήχο των, της κίνησης που ξεπερνά τα 55 δεσιπέλ. Σε όλη την Ευρώπη σχεδόν ένας στους δύο υποφέρει από τον θόρυβο της κίνησης. Έχουμε πρόορους θανάτους, 50.000 λόγω αυτού αναφέρουν ε, τα στοιχεία και από 2.000 μέχρι 50.000 καρδιακές προσβολές. Άλλα προβλήματα είναι η ψυχική υγεία και η έλλειψη ύπνου, κάτι το οποίο αυξάνει και το κίνδυνο ε, εμφάνισης διαβήτη και άλλων νοσημάτων. Το πιο απλό είναι να μειωθεί το επίπεδο θορύβου στο όχημα αυτό καθεαυτό. Αυτό, αυτό ζητούν ε, και οι καταναλωτές περισσότερο η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη. Ένα ε, στα τρία οχήματα και ένα στα τρία φορτηγά εκπληρώνει τις προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή. Με την, στην Επιτροπή ΕΜΒΗ η συμβαστική λύση που επιτεύχθηκε εκεί θα μετριάσει ακόμα περισσότερο την πρόταση της Επιτροπής. Οι πράσινοι δέχθηκαν δεν δέχτηκα να προχωρήσει αυτή η τόσο αποδυναμωμένη πρόταση από το ΕΛΚΑ. Σίγουρα βέβαια το όφελος ξεπερνάει το κόστος κατά πολύ. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να στηρίξουν αυτή την άποψη. Σας ζητώ να στηρίξετε την τροπολογία 67 για μείωση ε, των δεσιμπέλ σε 10 χρόνια κατά 2 δεσιμπέλ. Εκπλήσωμαι διότι το ΕΛΚ υπέγραψε τρεις τρυπολογίες με τον ίδιο σκοπό. Νομίζω ότι αυτό δεν επιτρέπεται σε καμία άλλη πολιτική ομάδα και δεν ξέρω πώς έγινε εδώ. Ειδικότερα ως προς τη μείωση του κόστους του δημοσίου τομέα. Θα ήθελα να πω γι' αυτό ότι Πράγματι θα μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες ε, αν μειώσουμε και το κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Εάν θα έχουμε ε, φράγματα θορύβου αν τελικά αυτά κατασκευάσουμε στους αυτοκινητόδρομους, αυτό το κόστος θα επιβαρύνει πολύ ε, τους πολίτες και τα δημόσια οικονομικά. Είναι καλύτερο να μειωθεί ο θόρυβος στην πηγή οι διαχειριστές και οι μεγάλοι διευθυντές της αυτοκινητοβιομηχανίας μπορούν να ζήσουν και ζουν άλλωστε πολύ μακριά από εκεί όπου, σημειώνεται ο θόρυβος. Οι φτωχοί είναι που υποφέρουν περισσότερο. Ο κύριος Μπάτεν. Η, η έκθεση αυτή προτείνει τη μείωση του θορύβου της ηχοστάθμης των μηχανοκίνητων οχημάτων και θα επιφέρει ε, περισσότερη γραφειοκρατία. Αναφέρει η έκθεση ότι η ποιότητα του οδοστρώματος ίσως είναι η λύση στο πρόβλημα. Ίσως, αλλά πόσο θα στοιχήσει και έτσι όπως έχουν τα οικονομικά των κρατών μελών, πού θα βρεθούν τα χρήματα για να ε, γίνει αυτό το κολοσιαίο έργο. Και αν είναι κανονισμός θα έχει άμεση αυτόματη νομικός δεσμευτική ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη και οι δημοκρατικώς εκλεγμένες εθνικές κυβερνήσεις δεν θα έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν αν θα θέλουν να εφαρμόσουν τον κανονισμό ή όχι. Δεν έχουν επιλογή, οφείλουν να τον εφαρμόσουν. Ίσως είναι μία από αυτές τις εξουσίες και αρμοδιότητες που θέλει ο Ντέβιτ Κάμερον να επαναδιαπραγματευτεί για να επιστρέψει ως αρμοδιότητα στο ε, Βρετανικό Κοινοβούλιο. Μέχρι ότου τα καταφέρει θα πρέπει να συνεχίσει να ε, υποκύπτει στους αφέντες του στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ για δύο λεπτά η κυρία Βίλς. Ευχαριστώ πολύ. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας του ΟΗΕ υπολόγισε τις επιπτώσεις ε, του θορύβου στην ανθρώπινη υγεία. Μετά την ατμοσφαιρική ρήπανση, ο θόρυβος είναι ο πιο επιβαρυντικός για την υγεία. Περίπου 210 εκατομμύρια πολίτες ε, στην Ένωση εκτίθεται σε θόρυβο πάνω από 55 δεσιπέλ και πολλοί εξ αυτών και τη νύχτα. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην ακοή, στον ύπνο, ε, στρες, καρδιακά νοσήματα και ε, προβλήματα στα παιδιά. Και παρακαλώ, δεν θα πρέπει να το υποτιμούμε αυτό. Ακόμα και μικρή μείωση όμως του θορύβου μπορεί να έχει μεγάλα αποτελέσματα. Γιατί από το 1992 δεν έχουν αλλάξει οι οριακές τιμές για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πρόταση. Το αποτέλεσμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα πρέπει να το διατηρήσουμε με τις νέες οριακές τιμές. Ήδη από σήμερα συμμορφώνονται ορισμένα οχήματα. Ε, γιατί όμως τίθενται σε ισχύ οι νέες τιμές μετά από μία επταετία. Θα περιμένουμε να προσαρμοστούν ε, όλες οι εταιρείες, η τεχνολογία υπάρχει από σήμερα. Μέχρι τώρα η νομοθετική διαδικασία έχει δείξει ότι ο νέος κανονισμός ε, υποφέρει μαζικά από την πίεση των λόμπι. Η αυτοκίνητο βιομηχανία και οι σύνδεσμοί της υποτιμούν ε, το θόρυβο, εμποδίζει νέες έρευνες και νέους υπολογισμούς τους χαρακτηρίζει μη σοβαρούς. Για ποιο λόγο Εδώ και δεκαετίε μιλούμε γιατί δεν υπολογίζουν, δεν συνυπολογίζουν στο κόστος τους οι αυτοκινητοβιομηχανίε τον παράγοντα πληθωρισμό. Θέλουν να μετακυλήσουν το κόστος στους καταναλωτέ για να μειωθεί ο θόρυβο στα αυτοκίνητα που παράγουν. Ευχαριστώ για ένα λεπτό η κυρία Σόσα Βάγνερ. Ο κύριο Σόσα Βάγνερ, διορθώνει πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από τότε που είμαι εγώ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχω ξεκινήσει μια μικρή σταυροφορία κατά του θορύβου που παράγουν ε, οι μηχανές ε, με τις λεγόμενες ε, πειραγμένες εξατμίσεις. Και θα πρέπει να δούμε πώς πάσχει ο πληθυσμός από τους θορύβους αυτούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μου έδισαν οι ειδικοί, είναι τεχνικός δυνατόν για τους ε, κατασκευαστές μηχανών να μειώσουν ή να περιορίσουν αυτές τις ε, ε, εξατμίσεις. Εξακολουθεί βέβαια να μην εισακούγεται στην ομοθεσία η έκκλησή μου. Ε, με την ομοθεσία αυτή την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία πραγματικά είναι ε, χαόδης. Για δύο λεπτά ο κύριος Ζήμπερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι ο θόρυβος είναι ένα πρόβλημα και για την υγεία των ανθρώπων και για το περιβάλλον. Είναι πολλές οι μελέτες ε, και οι ποοί υπολογίζει ε, σε ένα εκατομμύριο τα ε, έτη υγιού ζωής που χάνουν οι Ευρωπαίοι κάθε χρόνο. Για μένα είναι σημαντικό να δούμε το συνολικό πρόβλημα και τη στρατηγική και να μην το περιορίζουμε σε κινητήρες ή σε μείωση του θορύβου με σιγαστήρες ας πούμε ε, τα ελαστικά, την αεροδυναμική, ε, το δόστρωμα. Ε, είναι ένα γενικό θέμα ο θόρυβος, δεν είναι μεμονωμένη πηγή θορύβου, δεν φταίει ένα μόνο στοιχείο. Τώρα θα πρέπει να κοιτάξουμε, αφού συζητούμε το κανονισμό αυτό, να καταλάβουμε ότι κάθε αυτοκίνητο ξεχωριστά θα πρέπει να ε, εφαρμόζει και να τηρεί αυτές τις προδιαγραφές και ε, όχι ε, όπως ισχύει με το διοξίδι του άνθρακα που αφορά όλο το στόλο των οχημάτων. Θα πρέπει να υπολογίσουμε λοιπόν το κόστος και αν ισχύσουν ε, για τον κινητήρα αυτές οι ρυθμίσεις θα σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα θα γίνουν και πιο βαριά άρα και πιο ακριβά. Έτσι να το έχουμε υπόψη μας. Τι μας ενοχλεί εμάς στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπόθηκε προηγουμένως, ε, είναι το παράρτημα 3 και η παλιά ταξινόμηση. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Και γι' αυτό η νομοθετική διαδικασία διήρκησε τόσο πολύ γιατί χρειάστηκε να διορθωθούν όλα αυτά. Με τη δική μας λοιπόν τροπολογία 61 προσπαθήσαμε ε, βάσει της σύστασης του ΙΕ να κατατάξουμε σωστά και ρεαλιστικά ε, τα οχήματα. Ευτυχώς ε, ε, και αυτό δεν είναι πλέον επίμαχο. για να προστατεύουμε και άτομα με αναπηρία από οχήματα που πλέον δεν θα μπορούν να αντιλαμβάνονται γιατί θα είναι τόσο αθόρυβα. Ευχαριστώ για δύο λεπτά ο κύριος Γκρότερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι από τον Επίτροπο Υγείας, ούτε από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, αλλά από τον Επίτροπο Βιομηχανίας. Και ακούω για την πτώση και την παρακμή και το τέλος της αυτοκινητοβιομηχανίας και εκπλήσωμαι πάρα πολύ. Η πρόταση είναι λογική. Στη βάση της ε, θα πρέπει να σφυριλατήσουμε ένα συμβασμό εγώ ενοχλούμε γιατί πρέπει να γίνει σε πρώτη ανάγνωση και ο χρόνος που χρειαστήκαν ε, να αντιμετωπίσουμε και να διεκπαιρεώσουμε την έκθεση δεν έχει να κάνει με δική μας ολιγορία. Υπήρχαν προβλήματα. Για να δούμε ε, πού είναι τα ελλείμματα, ποιες είναι οι επιρροές που ασκούνται, γι' αυτό χρειάστηκε τόσο καιρό. Ο κάθε άνθρωπος μια ζωή έχει και μια υγεία την έχει. Θα πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Να μειωθούν οι πηγές ενόχλησης. Ε, δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα πάντα. Το δόστρωμα είναι υπόθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι και οι κοινότητες τα κάνουν αυτά στα κράτη-μέλη. Κάτω τα χέρια. Τι δουλειά έχουμε να κατεβόμαστε εκεί. Έχουμε ε, ένα πεδίο αρμοδιοτήτων δεδομένο και γνωστό. Γι' αυτό στην Επιτροπή Περιβάλλοντος νομίζω ε, καταλήξαμε σε μια καλή επιλογή και βρισκόμαστε αγαπητοί συνάδελφοι στην αρχή των διαπραγματεύσεων. Πρώτη ανάγνωση. Γιατί να βιαζόμαστε. 60 70% ε, στο περιβάλλον ε, έχει διεκπαιρεωθεί σε πρώτη ανάγνωση. Είναι και θέμα δημοκρατίας για τέτοια πράγματα που έχουν τεράστιες επιπτώσεις και στην υγεία και στη βιομηχανία. Μήπως χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο κανονική δεύτερη ανάγνωση. Με την ησυχία μας να συμμετέχουν όλοι και εκτός του Κοινοβουλίου ενδιαφερόμενοι για να διαμορφώσουν άποψη. Σε πρώτη ανάγνωση αυτό δεν είναι δεδομένο άρον άρον το περνάμε. Αυτό θέλω να το ε, καταδείξω και να μην υποχωρήσουμε πίσω από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι αυτή η κόκκινη γραμμή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάντερς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε οι μεταφορές, οι οδικές μεταφορές, τα αυτοκίνητα μας έχουν φέρει μεγάλη ευημερία και θέση εργασίας, πολύ ωραία, αλλά και η κυκλοφορία δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα με το θόρυβο, το συζητούμε. Και ε, σε συνεργασία με τη βιομηχανία θα πρέπει να υποχωρήσει. Ε, αν συμφωνήσει η βιομηχανία δεν χρειάζεται το κόστος να το επιμίζεται ε, μόνο το δημόσιο. Ε, φτιάχνουμε διάφορα φράγματα, ε, ε, ηχομονώσεις και τέτοια στους αυτοκινητοδρόμους. Καλά κάνουμε, αλλά θα πρέπει και η βιομηχανία να αναλάβει τις ευθύνες της. Ε, νομίζω ότι είναι ισόρροπη η πρόταση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, στην Ευρώπη ελπίζω να έχουμε και όλες τις μεθόδους ε, τεστ και δοκιμών για να μετράμε τα ίδια πράγματα. Και τελικά να είναι και καλύτερη η ανταγωνιστική θέση της Ευρωπαϊκής Αυτοκινητομηχανίας, Πρόεδρε, γιατί η τεχνική πρόοδος είναι πλεονέκτημα ανταγωνιστικό σε αυτά τα θέματα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για δύο λεπτά ο κύριος Εκχάουτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κλασική συζήτηση, απίστευτα κλασική. Βρίσκουμε ένα θέμα, ε, ωραία, ε, ε, θόρυβος που ενοχλεί πολύ κόσμο και τι να κάνουμε. Και πρέπει να το κάνει η Ευρώπη για να υπάρχει για όλους τους κατασκευαστές το ίδιο γήπεδο, με τους ίδιους κανόνες. Ωραία βρέπουμε ένα θέμα και μας λένε οι συντηρητικοί «Α, όχι, είναι πολύ ακριβό για τους ε, κατασκευαστές, η κρίση δεν έχει περάσει ακόμα, σιγά-σιγά». Και ξαφνικά δεν μιλάνε για το κόστος που πληρώνει η κοινωνία για να χτίζουμε αυτά τα φράγματα τα ηχομονωτικά ή ο κόσμος που υποφέρει από το θόρυβο. Αυτό δεν το συζητάμε. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τι πρέπει να κάνει η βιομηχανία για να προσαρμοστεί με την καινοτομία για να μπορεί να είναι διεθνώς πιο ανταγωνιστική. Και ξαφνικά έρχεται η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που από ό,τι φαίνεται είναι σούπερ φιλόδοξη. περίεργο αυτό. Τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, υπερεύει αυτόν. Τι είναι αυτά που κάνετε, ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία ε, επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόμπι. Είναι μια πρόταση που σημαίνει λιγότερο θόρυβο, λιγότερη επιβάρυνση ε, για ε, την κοινωνία και ε, για την υγεία. Γι' αυτό είμαι κατά της ε, τροπολογίας 61 που θέλει να αποδυναμώσει την πρόταση. Εμείς παραμένουμε ε, στην πρόταση της τροπολογίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και να μην είμαστε η φωνή της αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι πολύ ε, σφριγγυλή και ζωντανή ακόμα η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη και δεν έχει ανάγκη. Ευχαριστώ για δύο λεπτά κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι εδώ πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας της υγείας και της επιμερίας των καταναλωτών από τη μία αλλά και από την άλλη τη δυνατότητα ανταγωνιστικότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το πρόβλημα με την έκθεση αυτή είναι το παράρτημα 3 με το κατόφλι που προτείνει η κυρία Μέρκης ένα κατόφλι που δεν συνάδει ούτε με την τεχνική λογική ούτε με την επιστημονική λογική. Όταν μιλούμε για σιωπηλό κινητήρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την πρόσβηση με το έδαφος, ε, το είδος της ασφαλτόστρωσης το δόστρωμα, αλλά και την κατάσταση των ελαστικών. Βεβαίως δεν μπορούν να τα ελέγξουν όλα αυτά οι κατασκευαστές των αυτοκινήτων των αυτοκινήτων, αλλά είναι προτιμότερο να τους ζητήσουμε να προοδεύσουν σε αυτό το τομέα αναστάδια, σιγά σιγά. Εν πάση περιπτώσει να μην τους στραγγαλίσουμε εξαναγκάσοντάς τους πάρα πολύ γρήγορα να πετύχουν κατόφλια τα οποία τελικά δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Άλλωστε, ως προς τα ελαστικά των αυτοκινήτων θα πρέπει οι δοκιμές να μην γίνονται με καινούρια λάστιχα αλλά να γίνονται στις πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας όπου έχουμε ε, ελαστικά σε διάφορες καταστάσεις, πολλές και διαφορετικές. Εμείς είμαστε κατά της τροπολογίας 68 και βεβαίως της τροπολογίας 51 διότι πάνε υπερβολικά μακριά. Είναι σημαντικό κατά την άποψή μου στην υπόθεση αυτή να ξέρουμε ποια είναι η αποστολή μας έναντι των εκλογέων μας. Είναι δύσκολη η περίοδος και θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Από τη μία να προστατεύσουμε την υγεία, από την άλλη να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος Πυρίλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η χορύπανση και οι συνέπειές της στην ανθρώπινη υγεία δεν θα πρέπει να υποτιμούνται. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να ε, μειώσουμε το επίπεδο θορύβου των αυτοκινήτων οχημάτων που προτείνονται στο συγκεκριμένο κανονισμό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις οικονομικές ε, προσπάθειες που απαιτούνται από πλευρά της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ε, Ένα κλάδο ο οποίο είναι στρατηγική σημασία για τη δημιουργία θέσεων εργασίων που πλήττεται αυτή τη στιγμή από την κρίση. Αυτά τα οποία προτείνονται στο παράρτημα 3 φαίνεται να μην είναι ρεαλιστική φύσεω και όσον αφορά την τεχνολογία και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει να αποφύγουμε να υπάρχει υπερβολική ρύθμιση για τον τομέα. Εγώ είμαι υπέρ τη ε, διάταξη άβαση, η οποία λαμβάνει υπόψη και κάποιε κατηγορίε ανθρώπων που πρέπει να προστατεύονται, όπω για παράδειγμα τα παιδιά και οι τυφλοί, οι οποίοι κινδυνεύουν από ηλεκτρικά οχήματα, επί παραδείγματα, που έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Η κυρία Σάβισαρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η μείωση των επιπέδων θορύβου είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους κατασκευαστές ε, λαφρεών και βαρέων οχημάτων. Στην περίπτωση των βαρέων οχημάτων, ε, το βασικό πρόβλημα είναι η ταξινόμηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει δύο κατηγορίες ταξινόμησης, αλλά επαρκεί αυτό. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και πού πηγαίνουν αυτά τα οχήματα και τι μεταφέρουν και ε, τι γίνεται και με τις μεταφορικές εταιρείες για να δημιουργήσουμε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα ε, κάτω από 80, 180, 180 με 500 ε, και πάνω από 500. Αυτό θα μας διασφαλίσει ότι θα έχουμε ομαλή ε, μεταφορά μεγάλων όγκων αγαθών. Και αυτό φυσικά σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε και ανάλογα επίπεδα ασφαλείας για μεγάλα λεωφορεία. Υπάρχουν και κάποια προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή ε, για τα κατάλληλα επίπεδα θορύβου. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα μπορεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις εντός των ε, προθεσμιών. Και θα πρέπει οι προσπάθειές μας να συμβαδίζουν και με την ενίσχυση του μεταφορικού τομέα. Ελπίζω να έχουμε μια ισορροπημένη πρόταση. Για δύο λεπτά η κυρία Μουρκουνάιτε Μικουλένιενε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. τέτοια ώρα νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλάμε για επίπεδα θορύβου. Όσο λιγότερος ο θόρυβος, τόσο καλύτερα θα κοιμηθούμε. Δύο θέματα θα ήθελα να θίξω. Καταρχάς, ε, οι δοκιμές ε, MOT που θα πρέπει να διεξάγουν οι χώρες μέλη υπάρχει μια συνολική βάση έγκρισης ταξινόμησης που περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες εκπομπές θορύβου. Από ό,τι φαίνεται όμω, κάποια κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν τα βάση ε, δεδομένων αυτήν όταν κάνουν τι κατάλληλε δοκιμίε, αλλά υπολογίζουν τα επίπεδα του θορύβου με βάση ε, τα παραμέτρου του κινητήρα. Είναι παροχημένε αυτέ οι μέθοδοι και αποδεικνύεται ότι υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν ακόμα στου δρόμου και παράγουν ε, θορύβους που είναι επιζήμιοι για την υγεία μα. Ε, στην περίπτωση των μεταχειρισμένων οχημάτων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ηλικία του οχήματο. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται καμία παρέκκληση στα επίπεδα θορύβου που καθορίζονται από του ευρωπαϊκού κανόνε. Ε, θα ήθελα επίσης να σταθώ στις αρνητικές συνέπειες ε, του στόχου που έχουμε εδώ στη συγκεκριμένη πρόταση. Θέλουμε να μειώσουμε τα επίπεδα θορύβου των οχημάτων ακούστηκε επανειλημμένο και θα το επαναλάβω κι εγώ. Η απουσία θορύβου στα ηλεκτρικά οχήματα θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ε, ε, τυφλών ατόμων και γι' αυτό ακριβώς ε, τα οχήματα αυτά θα πρέπει να έχουν συστήματα ήχου τα οποία να επιτρέπουν να τα εντοπίζουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. λέει κύριε Βέστλον. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το θέμα αυτό. Πρέπει να ληφθούν μέτρα, τα οποία σίγουρα θα στοιχήσουν. Και πολύ συχνά στοιχίζουν ακριβά αυτά τα μέτρα. Αυτό είναι αληθές. Και η αυτοκινητοβιομηχανία περνάει δύσκολες στιγμές. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Και αντιμετωπίζει μια πολύ μεγάλη πρόκληση θέλει να υιοθετήσει πιο οικολογικές τεχνολογίες με μικρότερη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Από την άλλη έχει πολύ μακρά περίοδο παραγωγικής διαδικασίας, ειδικά ως προς τα βαρέα οχήματα, αλλά και ως προς τα πιο ελαφριά οχήματα. Σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο κύριος Περέγιο Ροντρίγκεθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να έχουμε την ετοιμότητα να αναγνωρίσουμε ότι η πολιτική για την αντιμετώπιση της ε, χορύπανσης ε, είναι κρεμίσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίποτα δεν έχει γίνει και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όταν θα ψηφίσουμε. Όταν ε, ασχοληθήκαμε με την έκθεση για τα αεροπλάνα, εγώ προσωπικά γνώρισα ανθρώπους που έχουν πληγεί. Η υγεία τους έχει πληγεί από τα επίπεδα θορύβου. Η Επιτροπή παρουσιάζει μια πολύ καλή πρόταση στην με την έκθεση αυτή, με το παράρτημα 3. Όσοι νομίζουν ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξη η πρόταση αυτή, να ξέρουν ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα για την επίτευξη σωστή ισορροπίας μεταξύ του προστατευτισμού του Συμβουλίου και των φιλοδοξιών του Κοινοβουλίου. Εάν θεωρήσουμε ότι είναι σοβαρή η έκθεση αντικτύπου της Επιτροπής, τότε ή ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι αλήθεια ότι θα υπάρξει αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας. Μιλούμε για την ηχορύμπανση και δεν μιλούμε για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Τους καλώ όλους λοιπόν τους συναδέλφου να, το, να την υπερψηφίσουν την έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Φαν Μπρέμπτ. Συνάδελφοι. Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού στην Ευρώπη σήμερα ζει στις πόλεις και θα αυξηθεί αυτό. Πρέπει να βρούμε μια λύση και για το κλίμα και για τη χωροταξία και ε, για την εγκύτητα στις πόλεις θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να λύσουμε κάποια ε, δύσκολα ε, προβλήματα στις πόλεις. Στην πόλη μου την Αμβέρσα δείχνει μια πρόσφατη μελέτη ότι ένα στους δύο κατοίκους ενοχλείται από το θόρυβο και μάλιστα από επίμονο θόρυβο με προβλήματα και υγείας που ανέφερε ο Επίτροπος. Ε, είναι οπωσδήποτε καθήκον μας να το αντιμετωπίσουμε. Δεν έχει νόημα να συζητάμε ε, για τα προβλήματα που υπάρχουν στην αυτοκινητομηχανία που τα ξέρω γιατί και στη δική μου πόλη έχω τέτοια στη γειτονιά μου. Θα πρέπει να δούμε, ξέρω εγώ, να προσαρμόζεται το οδόστρωμα ή άσφαλτος, να φτιάχνουμε φράγματα στους αυτοκινητοδρόμους, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ε, και έχουμε επιτύχει ένα συμβιβασμό με ε, μεγάλη προσπάθεια στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα πρέπει και η δεξιά πλευρά του Κοινοβουλίου να τον τηρήσει. Ο κύριος Λιμπεράτσκι, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, άκουσα τους διάφορους ομιλητές και νομίζω ότι είναι μάλλον μετριοπαθής η πρόταση τα οχήματα μπορεί να εκπέμπουν μέχρι 80 δεσιμπέλ και εμείς θέλουμε να μειώσουμε μερικά δεσιμπέλ. Δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αυτό για την αυτοκινητοβιομηχανία. Εάν ε, ο κινητήρας στοιχίζει περισσότερο, τότε θα δαπανούμε λιγότερα σε ηχοφράγματα. και με ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονό ότι θέλει να λάβει μέτρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για του αυτοκινητοδρόμου ε, και τη μείωση του θορύβου των οχημάτων. Όλα αυτά αναφέρονται στο παράρτημα 3 στην πρόταση του εισηγητή δεν θεωρώ ότι είναι η καλύτερη δυνατή λύση η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αρχική πρόταση στο παράρτημα 3, ε, η πρόταση του εισηγητή, η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν καλύτερη. Μας επέτρεπε να ε, κατασκευάσουμε καλύτερα αυτοκινήτα τα οποία είναι τα λιλότερα για τους πολίτες μας και για την υγεία τους. Ωραία, θα ολοκληρώσουμε τώρα τη συζήτηση με τη διαδικασία του ΚΑΤΣΔΙ. Η κυρία Μπασέσκου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι μία από τις βασικές πηγές θορύβου είναι η οδική μεταφορά. Έχουμε διαταραχές ύπνου, έχουμε καρδιακές διαταραχές, έχουμε ε, προβλήματα στην ε, εγκεφαλική λειτουργία. Όλα αυτά ε, προκύπτουν από μεγάλη έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου. Είναι σαφέστατος ο αρνητικός αντίκτυπος της συγχωρήπανσης και στην υγεία αλλά και στο περιβάλλον. Η Ντάτσια που ανήκει στη Ρενό είναι μεγάλος κατασκευαστής στην αυτοκινητοβιομηχανία τα τελευταία χρόνια. Ε, ανήκει στη χώρα μου τη Ρουμανία και ενδεχομένως γι' αυτό η κυβέρνηση, ε, η χώρα μου δεν έχει κινηθεί σωστά προς αυτή την κατεύθυνση μερικές φορές. Νομίζω ότι οι καταναλωτές χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, να έχουμε διαφάνεια στα στοιχεία ως προς τα επίπεδα θορύβου για να, έχουν, να μπορούν ενημερωμένα να πάρουν τις αποφάσεις τους. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, 80% του πληθυσμού ζει στις πόλεις και σύμφωνα με ειδικούς για το περιβάλλον ο θόρυβος είναι υπερβολικός στις πόλεις. Θα πρέπει ε, με τις νέες τεχνολογίες, ε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ε, να ε, προσαρμοστούμε. Αλλά τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι σχεδόν αθόρυβα και ε, είναι απειλή για τους τυφλούς ή για κάποιους απρόσεκτους πεζούς. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα προειδοποίησης με ένα ηχητικό σήμα. Ε, αντίστοιχο με κάποιες ε, σημάσεις που υπάρχουν σε φανάρια ή σε σιδηροδρομικές διαβάσεις για να ειδοποιούνται οι πεζοί. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα προειδοποίησης ε, για να αποφεύγονται τα οδικά δυστυχήματα. Και ε, τώρα ήρθε η ώρα να ολοκληρώσει ο Επίτροπος κ. Σταγιάννη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εχθέ το βράδυ επανέλαβα ότι είναι πολύ σημαντικό από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά και από πλευρά μου που είμαι αρμόδιο για την ε, βιομηχανική πολιτική, να ξεκινήσουμε μια διαδικασία για την ε, εκ νέου εκβιομηχανιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια σαφή επιλογή μας Αλλά η βιομηχανική ε, ε, πολιτική που έχω εγώ κατά νου θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια βιομηχανία που Πόρα απέχει από τη βιομηχανία της δεκαετίας ε, του 80 και του 90. Θα πρέπει να είναι μια σύγχρονη βιομηχανία, ανταγωνιστική, υψηλού επίπεδου, που θα πρωταγωνιστεί στην πράσινη οικονομία. Και επομένως θα πρωταγωνιστεί και στις δράσεις μας ε, στην, ε, για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος μια ισορροπημένη πολιτική βεβαίως όπου η πολιτική ε, για την υγεία και η βιομηχανική πολιτική θα μπορούν να συνεργάζονται και να έχουν όλες ένα κοινό στόχο, να ζουν καλύτερα οι πολίτες μας. Η πρότασή μου, και εδώ θα ήθελα να καθησυχάσω την κυρία Γκροστέτ και τον κύριο Ταταρέλα, σαφώς δεν είναι μια πρόταση κατά της βιομηχανίας, ιδίως κατά της αυτοβιομηχανίας. Στο έγγραφο που αναφέρεται στην πολιτική υπέρ της βιομηχανοποίησης της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί ένα από του ζωτικού τομεί. Αλλά εμεί έχουμε κατά νου ένα πιο οικολογικό αυτοκίνητο που θα ρηπαίνει λιγότερο, όχι μόνο όσον αφορά τις εκπομπές διοξίδιου του άνθρακα, αλλά και όσον αφορά την ηχορύπανση. Και η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την άποψή μου, είναι μια πρόταση που προσπαθεί να συγκεράσει τα διάφορα συμφέροντα. Βιομηχανική πολιτική και προστασία τη αυτοβιομηχανία. Δεν υπάρχουν υπερβολή στην πρόταση, δεν είναι ακραία πρόταση, αλλά είναι μια μια πρόταση που προσπαθεί να προστατεύσει μια σύγχρονη και ανταγωνιστική βιομηχανία και ταυτόχρονα και το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι καθόλου διατεθειμένος να εξετάσω τροπολογίες οι οποίες βελτιώνουν το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα. Και στη διάρκεια της συζήτησης και στη συνέχεια και της ψηφοφορία στο Συμβούλιο και στη συζήτηση στο Συμβούλιο είμαστε, όπως σας είπα, καθόλου διατεθειμένοι να συνεργαστούμε προκειμένου το κείμενο του νέου κανονισμού να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο πρέπει να πω ότι πολλά από αυτά τα οποία ζητούμε για κάποια οχήματα ισχύουν ήδη υπό την έννοια ότι ε, συμμορφούνται προς την νομοθεσία που προτείνουμε. Γι' αυτό ακριβώς ε, και για κάποιες άλλες περιπτώσεις ε, ε, για την πρώτη περίπτωση να μην είναι εύκολα, αλλά το δεύτερο στάδιο για την περαιτέρω μείωση θα είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι είναι επαρκής χρόνος αυτός ο οποίος δίνεται, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα η αυτοκινητοβιομηχανία. Αλλά από πλευράς αποσχόλησης δεν νομίζω ότι ο συγκεκριμένο κανονισμός θα προκαλέσει ζημία. Ίσα ίσα, κατά την άποψή μου, μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει μια βιομηχανία που θα είναι πιο ανταγωνιστική. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι η συγκεκριμένη πρόταση κανονισμού είναι ισορροπημένη και επιβεβαιώνω παρόλα αυτά ότι είμαι καθόλου διατεθειμένος να συνεργαστώ μαζί σας από σήμερα και για τους επόμενους μήνες μέχρι να εγκριθεί η πρόταση από το Συμβούλιο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα είναι ισορροπημένο και θα είναι προς το συμφέρον των πολιτών μας. Διότι εμείς πιστεύουμε σίγουρα στην αγορά, πιστεύουμε στη βιομηχανία, αλλά Όλα αυτά αποτελούν εργαλείο και ως τελικό στόχο έχουμε, και θα το επαναλαμβάνω συνεχώς, την κοινωνική πολιτική. Δηλαδή να βοηθήσουμε τους πολίτες μας να ζουν καλύτερα και όσον αφορά την υγεία τους και όσον αφορά τις οικονομικές τους ε, δυνατότητες. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τους βουλευτές ε, που είπαν ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι και μάλλον και παραπάνω φιλόδοξη από όσο πρέπει. Ε, και χθε άκουσα σε μια άλλη συζήτηση ε, καλά λόγια για τις προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι η αίσθηση ε, και η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ολομέλειας εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος. Τελευταίος για σήμερα ο εισηγητής ο κύριος Μύροσλαβ Όσκι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές ε, για τη συνεισφορά τους. Η συζήτηση πραγματικά ήταν ε, μια καλή εικόνα των συζητήσεων που είχαμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ε, το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι όλη αυτή η νομοθεσία εντάσσεται στο πλαίσιο των θεμάτων του θορύβου που είναι πάρα πολύ φλέγοντα. Και όλα αυτά τα θέματα χρειάζονται καλύτερη αξιολόγηση από πλευράς των ειδικών και των εμπειρογνωμόνων. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα αυτά που είπατε, γιατί όταν είσαι πολιτικός δεν μπορείς να ασχολείσαι με δεσιμπέλ, ένα δεσιμπέλ πάνω, ένα δεσιμπέλ κάτω, αλλάζει, είναι αποφασιστικό. Αυτά εμείς δεν τα ξέρουμε, αλλά θα ήθελα να απαντήσω ε, σε εκείνα τα σχόλια που αναφέρθηκαν σε ε, απειλές, ε, ότι συνιστά αυτό απειλή δηλαδή για την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Εμείς θεωρούμε ότι δεν ευσταθεί αυτό αν θεωρείτε ότι είναι απειλή. Πολύ συχνά ακούμε ότι η φιλόδοξη νομοθεσία μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης, εργασίας μάλλον. Ε, αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, αυτό μας απασχολεί και όταν νομοθετούμε. Το είπε και ο Επίτροπος. Πολύ συχνά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και πολύ συχνά με ρωτούν και πώ θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία με την παρούσα νομοθεσία. Με αν δούμε τι στατιστικές του κλάδου θα διαπιστώσουμε ότι μειώνονται οι πωλήσει, πέφτουν δυστυχώς στην Ευρώπη και θα πρέπει να κάνουμε κάτι ε, για το θόρυβο. Ας προσπαθήσουμε όσο μπορούμε για να μπορεί το Κοινοβούλιο να αποφανθεί και να συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο όσο γίνεται. Ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρία λέει ο Πρόεδρος. Ε, αύριο το πρωί επόμενη συνεδρίαση από τις 9 μέχρι τη 1 και το απόγευμα